από επιτυχία, από έναν προϋπολογισμό δηλαδή, στον οποίο όλοι θα συμφωνήσουμε. Thank you all. That item is now closed. Σας ευχαριστώ όλους. Πέρας του συγκεκριμένου θέματος. Περνάμε τώρα στο χρόνο ερωτήσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ζητώ συγγνώμη γιατί έχουμε καθυστερήσει λίγο. Αλλά στις 8.30 μέχρι τις 8.30 θα συνεχίσουμε. Θα ξεκινήσουμε με τις κατά προτεραιότητα χαρακτηρισμένες ερωτήσεις. Η πρώτη είναι η ερώτηση Παλέσκης. Μετά Elward, Μαγκίνες, μετά οι ερωτήσεις προς τους κυρίους κυρίους Άντορ, Πίλμπαγκς, ίσως έστω και μία ερώτηση για τον καθένα από αυτούς. Λυπάμαι γι' αυτό. Πρώτη ερώτηση λοιπόν είναι η 16. Ερώτηση υπαρίθμου 16. Για μια στιγμή. Μια στιγμή παρακαλώ. Για δικαστικό. Κύριο Μίτσελ, κοιτάξτε κανονικά έπρεπε να ξεκινήσουμε στις 7. Και η ερώτησή μου προς τον Επίτροπο για την Ανάπτυξη ε, δεν θα τη συζητήσουμε. Ίσως και να τη συζητήσουμε λέει ο Πρόεδρος. Όταν πήρα το Προεδρείο εδώ και αρκετή ώρα είχαμε μια καθυστέρηση μία ώρα. Τώρα έχουμε φτάσει σε μια καθυστέρηση μισή ώρα και προσπαθούμε να προλάβουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Λοιπόν, κύριε Ντεγκούχτο, να δώσετε απάντηση στην ερώτηση υπαρίθμου 16. Ερώτηση του κυρίου Παλέκης. Uh, uh, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μια ερώτηση που απαντώ εκ μέρους του Επιτρόπου Άτιγκερ και η απάντησή του είναι η εξής. Η δημόσια διαβούλευση που δημοσιεύθηκε στο, στο τόπο Voice in Europe το Μάιο Έλαβε 510 απαντήσεις ε, και πολλοί ενδιαφερόμενοι έστειλαν γραπτό σχόλια στη δημόσια διαβούλευση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με επιστολές και άλλες εκθέσεις. Σε γενικές γραμμέ, μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών της Ευρώπης είναι υπέρ δεσμευτικής κοινοτική νομοθεσίας από την οποία πολλοί αναμένουν ε, ενίσχυση των μέτρων ε, ασφάλειας και η έκθεση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής. Η νομοθετική πρόταση θα βασίζεται στο κεφάλαιο 3 της Συνθήκης Ευρατών που ασχολείται με θέματα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας. Στόχος είναι η δημιουργία ενός κοινοτικού πλαισίου για τα κράτη-μέλη που θα διασφαλίζει την ασφαλή διαχείριση καυσίμου και ραδιοενεργών αποβλήτων για όλα τα είδη των αποβλήτων σε όλα τα στάδια από τη δημιουργία μέχρι την ε, ε, συνεχίζονται οι συζητήσεις και είναι ακόμη πάρα πολύ νωρίς για να περιγράψουμε τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις θα παραμείνουν όμως αρμοδιότητα των κρατών μελών για τα ραδιενεργά απόβλητα. Ευχαριστώ. Κύριε Παλέτσκης, 30 δευτερόλεπτα επιπλέον. Mm, ačiū Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω για την απάντηση, η οποία όμως δεν ήταν και τόσο συγκεκριμένη. Εγώ πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να θέσει υψηλότερες περιβαλλοντικές απαιτήσεις στον τομέα αυτό. Θέλω λοιπόν να κάνω την εξή ερώτηση. Καταλαβαίνω ότι ο αρμόδιος επίτροπος για, την, για τον τομέα αυτό δεν παρίσταται. Θέλω όμως να σας ρωτήσω σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση των μέτρων αυτών θα υπάρχουν επαρκείς πόροι, επαρκή κονδύλια για να εξασφαλιστούμε ότι θα ληφθούν θετικέ για το περιβάλλον αποφάσεις. Ε, κυρία Τικάου, για μισό λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Η διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων και η αποθήκευσή του θα πρέπει να γίνεται σε συνθήκε μέγιστη ασφάλεια. Επομένω, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των εθνικών ε, περιφερειακών και τοπικών αρχών. Θέλω να ρωτήσω την Επιτροπή τι ρόλο βλέπει για τις τοπικές αρχές στη διαδικασία αυτή. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ντεχούχτα καλύπτει τον ε, κύριο Έτιγκερ. Δεν ξέρω αν θέλετε κύριε Έτιγκερ να... Μάλλον αν θέλετε, αν θέλετε κύριε Ντεχούχτα να απαντήσετε. Θα προσπαθήσω, λέει ο επίτροπο. Θα προσπαθήσω τουλάχιστον να μην πω ανοησίε. Σε ό,τι αφορά το πρώτο ερώτημα του κυρίου Παλέκη, η χρηματοδότηση, εξ όσων εγώ μπορώ να καταλάβω, είναι ένα θέμα, ε, πρόκειται για αρμοδιότητα των κρατών μελών. Το νομικό πλαίσιο είναι αυτό το οποίο θα θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκτιμώ λοιπόν ότι η χρηματοδότηση είναι εθνικό θέμα. Εκτός εάν στην νομοθεσία και από κοινού με τις δημοσιονομικές αρχές ληφθεί μια διαφορετική απόφαση. Εάν δεν συμβεί αυτό, ε, για τις τοπικές αρχές τώρα κυρία Τικάου νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με την ε, κατανομή εξουσιών ε, στο εκάστοτε κράτος μέλος. Εάν θα πρέπει οι τοπικές αρχές να δώσουν άδειε σε κάποιο βαθμό πράγματι θα είναι ένα μέρος της δικασίας λήψης αποφάσεων αλλά οι εγκρίσει ε, για κατασκευαστικά έργα, παραδείγματο χάρη, δίνονται σε εθνικό επίπεδο. Όλα αυτά θα τα δούμε στην νομοθεσία που θα σας προτείνουμε σύντομα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ντεχούχ τώρα για το ερώτημα 17 Έλγουτ. Έχετε το λόγο όταν είστε έτοιμος κύριε Επίτροπε. Ερώτηση 17. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η παιδική εργασία είναι κάτι το πάρα πολύ σοβαρό. Τον Ιούνιο το Διεθνές Γραφείο Εργασίας είπε ότι 240 εκατομμύρια παιδιά εργάζονται. Μειώνεται ο αριθμός των παιδιών αυτών βέβαια και αυτό είναι ενθαρρυντικό, αλλά παρόλα αυτά στον τρίτο κόσμο κυρίως τα παιδιά εργάζονται ενώ θα έπρεπε να μορφώνονται. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι μόνο το 5% των παιδιών αυτών εργάζονται σε τομείς εξαγωγικούς. Σύμφωνα με τα δεδομένα του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, τα περισσότερα παιδιά εργάζονται είτε σαν επιρρετικό προσωπικό είτε στη γεωργία για την παραγωγή τροφής. Προσπαθούμε να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα εκεί. Το πρόβλημα είναι προφανώς η φτώχεια και η έλλειψη εκπαίδευσης. Αυτό περιλαμβάνεται και στο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση της παιδικής εργασίας που έγινε δεκτό και από το Συμβούλιο της 14 Ιουνίου. Εκεί υπάρχουν πιο συγκεκριμένα στοιχεία για την πολιτική την οποία ακολουθούμε σχετικά με το πρόβλημα αυτό. Οι ενέργειές μας νομίζω ότι είναι συμβατές με τις διεθνείς προσπάθειες για την κατάργηση των χειρότερων μορφών παιδικής απασχόλησης μέχρι το 2014 πολλές ευρωπαϊκές εταιρείες, ακόμα και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στα πλαίσια των σχημάτων και των προγραμμάτων εταιρικής ευθύνης διασφαλίζουν το ότι δεν χρησιμοποιούνται παιδιά στην παραγωγή των προϊόντων τα οποία παράγουν ή εισάγουν. Και εξετάζει τα θέματα αυτά και στα πλαίσια της πολιτικής της Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, στις εταιρικέ σχέσεις με τις τρίτες χώρες. Έχουμε λοιπόν κάποια προγράμματα αηφορίες, τα οποία ελέγχουν τις εισαγωγές και την παραγωγή προϊόντων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα προγράμματα αυτά έτσι ώστε να μην χρησιμοποιείται ε, παιδική απασχόληση στα προϊόντα τα οποία τουλάχιστον εξάγονται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριος Aylward πρώτα, 30 δευτερόλεπτα. Κύριος Ρούμπικ μετά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτοί που ασχολούνται στην κοινωνία των πολιτών με το θέμα της παιδικής απασχόλησης θεωρούν ότι το θέμα αυτό πρέπει να χαρακτηρίζει τις αναπτυξιακές μας πολιτικές. Αν και το θέμα και από μόνο του έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Διαρωτώ με αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μια συγκεκριμένη πολιτική έτσι ώστε τα παιδιά αυτά τα οποία εργάζονται να επανέλθουν στην εκπαίδευση, στην παιδεία όπου τους χρειάζεται. Κύριε Επίτροπε, το ερώτημά μου αφορά τις διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ. Μπορεί στις διαπραγματεύσεις αυτές ε, να ξεκινήσει μια συζήτηση ε, για ένα σήμα ποιότητας ε, στο διεθνές εμπόριο ώστε ο καταναλωτής στην Ευρώπη να έχει την εγγύηση από ένα διεθνή οργανισμό, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, ότι αυτά τα προϊόντα έχουν παραχθεί χωρί να χρησιμοποιείται παιδική εργασία. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν κάτι που θα βοηθούσε ω μήνυμα που δίνουμε προ τα έξω. Ευχαριστώ. Κύριε Πίτρο, όταν ε, είστε έτοιμο, έχετε το λόγο. Με τη συμπληρω... Για τη συμπληρωματική ερώτηση του κ. Έλγουρτ θα ήθελα να προσθέσω ότι η τήρηση των συμβάσεων ε, τη Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας ε, για το θεμελιώδες ε, δικαίωμα στην εργασία. Αυτά αποτελούν ένα τμήμα και της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε σε πλαίσιο ρυθμίσεων γενικευμένων προτιμήσεων, είτε διμερών συμφωνιών. και σύμφωνα με τη διατάξει 138 και 182 για την παιδική εργασία και υπάρχουν και διατάξεις ε, για την ε, ε, τήρηση αυτών των διατάξεων και για το κοινωνικό διάλογο όπως υπάρχουν σε διάφορες εκθέσεις και συστάσεις. Η πολιτική μας δεν είναι το να αποσύρουμε προτιμήσεις ε, στο εμπόριο. Μπορούν να αποσυρθούν ε, τέτοιες προτιμησιακές συμφωνίες, μπορούμε να λάβουμε τέτοια μέτρα. Αλλά δεδομένου ότι μιλάμε για πολύ μικρό ποσοστό παιδιών ε, που εργάζονται σε επιχειρήσεις που είναι προσανατολισμένες προς τις εξαγωγές, η δράση μας θα έπρεπε μάλλον να είναι προληπτική και να έχουμε προγράμματα. Και έχουμε πολλά προγράμματα σε χώρες όπως η Ινδία, παραδείγματος χάρη, μέσω των οποίων φροντίζουμε για την ευημερία των παιδιών, ούτω ώστε να του διασφαλίζουμε και εκπαίδευση. Για το συμπληρωματικό ερώτημα για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει, θα ήθελα να πω ότι αυτά τα προγράμματα ακόμη και αν είναι οικειοθελή, μπορούν να προσθέσουν πολλά, αλλά όπω είπα και στην αρχική μου απάντηση, τα κράτη-μέλη πρέπει να, είναι, ε, να συμμετέχουν οικειοθελώ και είναι σίγουρο ότι η παιδική εργασία δεν μπορεί να αποτελέσει κομμάτι της ε, αλυσίδας ε, προσφοράς εργασίας. Ευχαριστώ πολύ και περνάμε στην ερώτηση 18 της κυρίας Μακίνες. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ανακοίνωση της 30 Ιουνίου για τη βελτίωση του συντονισμού, για τη σταθερότητα, την ανάπτυξη και τις απασχόληση, ουσιαστικά είναι η συνέχεια που είχαμε δώσει ε, στην ανακοίνηση. Θέλουμε ε, να παρουσιάσουμε συγκεκριμένα εργαλεία για το συντονισμό και προτείνουμε πιο αποτελεσματικό πλαίσιο επίβλεψης ε, και επιτήρησης, βελτιωμένη χρηματοοικονομική επιτήρηση, επιτήρηση των ανισοτήτων και ανισορροπιών και συντονισμό των οικονομικών πολιτικών. Στο πλαίσιο του οικονομικού εξαμήνου, προτάσεις μας έγιναν ε, ευνοϊκά δεκτές, υπάρχει ε, θετική αντίδραση και από την Task Force και από τα κράτη-μέλη και από τα μίδια στις 17 ε, Ιουνίου εγκρίθηκε η πρότασή μας και μας δόθηκε ενίσχυση να κάνουμε πραγματικότητα την καλύτερη οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρώπη το συντομότερο δυνατό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εγκρίνει τις απαραίτητες επίσημες προτάσεις εντός του τρέχοντος μήνα στο, ε, και βασιζόμαστε σίγουρα στη στήριξη από το Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο για να είναι όσο δυνατόν ε, πιο γρήγορα λειτουργικές αυτές οι προτάσεις. Θα προτείνουμε επίσης μια νέα εργαλειοθήκη κυρώσεων και ε, κινήτρων επίσης. Θα υπάρξουν επίσης μηχανισμοί ενίσχυσης για την εφαρμογή αυτών των φορολογικών κανόνων. Θέλουμε να είναι αξιόπιστο το φορολογικό πλαίσιο και αυτό είναι σημαντικό στοιχείο που συζητείται στην Task Force. Στην ανακοίνωση τη 30 Ιουνίου τονίζεται ότι θα προτείνουμε στην πρώτη φάση ένα νέο σύστημα κυρώσεων για τα 16 μέλη της Ευρωζώνης βάσει του άρθρου 136 της Συνθήκης Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε ό,τι αφορά το διορθωτικό ε, και προληπτικό και δεύτερον για το προληπτικό και το διορθωτικό σκέλος. Αυτά όλα δείχνουν ότι υπάρχει μεγαλύτερη αλληλεξάρτηση στη περίπτωση αυτή και θα υπάρχει συμπληρωματικότητα των κυρώσεων που προβλέπονται στο, σχέδιο, στο Σύμφωνο Σταθερότητας σε πιο πρόωρο στάδιο της διαδικασίας και με πιο αυτόματο τρόπο. Έπειτα θα υπάρχει το δεύτερο στάδιο που τα κράτη-μέλη θα μπορούν να προτείνουν την, ε, μπορούν την αναστολή κάποιων ε, πιστώσεων Παραδείγματο χάρη, κοινή πολιτική, πολιτική συνοχή και αλληλευτικό ταμείο. Στόχος μας θα είναι ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να είναι ένας επιπλέον μοχλός ε, άσκησης πίεσης για την τήρηση των απαιτήσεων ε, του συμφώνου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μαγκίνες και μετά κυρία Χάρκιν. Μισό λεπτό κυρία Μαγκίνες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή γιατί έδωσε μια ευρία απάντηση στην ανακοίνωση δεν διάβασα όλε αυτέ τι λεπτομέρειε, Βέβαια η ερώτησή μου είναι πιο συγκεκριμένη, γιατί υπάρχει η γνώση των πολιτών για, αυτές, για αυτές τις κυρώσεις. μπορείτε να τιμωρήσετε τι κυβερνήσει των κρατών μελών χωρίς να τιμωρήσετε του πολίτε, Ουσιαστικά αυτή είναι η ερώτησή μου. Εάν θέλετε να σταματήσετε τη ροή του προπολογισμού ε, στα κράτη-μέλη, στο πλαίσιο τη πολιτική συνοχή. Ε, Ποιο είναι αυτό ο οποίο ε, θα πληγεί και θα φυγεί από την περικοπή των πόρων. Αυτό θέλω να σα ρωτήσω. Κύριε Χάρκιν. Κύριε Επίτροπε, συμφωνώ ότι χρειάζονται κανόνε για την προστασία του κοινού νομίσματο. Όμω το Σύμφωνο Σταθερότητα ε, ε, προτάθηκε σε μια πολύ διαφορετική χρονική συγκυρία. Κάποιε χώρε τα καταφέρνουν καλύτερα από άλλε, οι δικοί μου και άλλε ε, παλεύουν, δυσκολεύονται. Το θέμα είναι ότι ε, όπως είπατε έχουμε δύο κατηγορίες κυρώσεων, όμως όπως και η κυρία Μαγκίνεσα αυτό θα πλήξει τους πολίτες. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι ο καλός τρόπος να συνεχίσουμε. Ξέρουμε ότι κάποιες χώρες βρίσκονται ακόμα στο χείλος της οικονομικής κατάρρευσης. Η Επιτροπή δεν νομίζω ότι προτείνει τα σωστά μέτρα. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπο, όταν είστε έτοιμος. Είμαι, είμαι έτοιμος. Ε, ακόμα και, και αυτή η ώρα κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι σημαντικό και τεχνικό ε, το ζήτημά σας ό,τι αφορά τα πολιετή προγράμματα. Η αναστολή των δημοσιονομικών δεσμεύσεων δεν θα επηρεάσουν ε, άμεσα τα πράγματα γιατί θα μπορούσαν να γίνουν οι πληρωμές. Και έχουμε έναν περίοδο διετίας για να προστατευθούν και κάποια projects και κάποια πολιετή προγράμματα. Και έτσι τα κράτη-μέλη θα έχουν ε, τον απαραίτητο χρόνο για να προβούν στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες. Τα ταμεία θα επαναγραφούν στον προπολογισμό, τα κονδύλια συγγνώμη, θα επαναγραφούν στον προπολογισμό όταν πλέον θα έχουν τηρήσει τα κράτη-μέλη τις υποχρεώσεις τους. Και οι κυρώσει επιβάλλονται μόνο όταν δεν έχει εκπληρώσει υποχρεώσει το κράτο μέλο. Και πάντω, σύμφωνα με την ανακοίνωση τη 30η Ιουνίου, από τον νέο μηχανισμό αποκλείονται καταστάσει όπου η μείωση δαπανών θα οδηγούσε σε μείωση του εισοδήματος αλλιέων και αγροτών. Σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό των κυρώσεων, εμείς έχουμε ως στόχο ακριβώς να εκπληρώσουμε τον όρο αυτό που σας προανέφερα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ντεχούχτ, ο Πρόεδρος, και για τη συντομία σας και για την σαφήνεια και ακρίβειά σας. Περνάμε τώρα στις ερωτήσεις προς τον κύριο Άντορ όταν είναι έτοιμος αρχής γενομένης με την ερώτηση παριθμών 19. Ερώτηση της κυρίας Μπλίνκεβιτσιούτε. Όπως προείπα αγαπητοί συνάδελφοι, δυστυχώς είμαστε πολύ πιεσμένοι σε ό,τι αφορά το χρόνο. Θα προσπαθήσω βέβαια να απαντηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες ερωτήσεις και θα παρακαλέσω να είστε όλοι σύντομοι. Ερώτηση 19. Άντορ. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι βουλευτές, Κατά την τελευταία δεκαετία υπήρξαν πολλές μεταρρυθμίσεις των συνταξιοδοτικών συστημάτων και συνεχίζονται στα κράτη-μέλη. Η Επιτροπή υποστηρίζει και παρακολουθεί και αξιολογεί την επίπτωση και την υλοποίηση των εθνικών μεταρρυθμίσεων με την ανοιχτή μέθοδο συντονισμού για να έχουμε τελικά συνταξιοδοτικά συστήματα που θα είναι και επαρκή και σύγχρονα και διαφανή η προσπάθεια παρακολούθησης και αξιολόγησης των συνταξιδοτικών συστημάτων περιλαμβάνει και την αξιολόγηση από την πολιτική οικονομικής πολιτικής και την Επιτροπή Πολιτικής Προστασίας. Λαμβάνουμε υπόψη τις διαργασίε των τελευταίων δέκα ετών μέσα στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης που καταλαβαίνουμε ότι αυτό δημιουργεί μια μεγαλύτερη πρόκληση για τις ε, συντάξεις ε, μέσα σε μια κοινωνία που γυράσκει και σε μια δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση. Το Συμβούλιο τον, ε, Ιούλιο, τον Ιούνιο υιοθέτησε μια διάμεση έκθεση και μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε μια συμπληρωματική έκθεση. Επίσης η Επιτροπή παρακολουθεί τις προσπάθειες των κρατών μελών σε πολλά συνταξιδοτικά προγράμματα. Υπάρχουν οι ετήσιες εκθέσεις και εκθέσεις ομοτήμων που αξιολογούν την κατάσταση στα μεμονωμένα κράτη-μέλη. Για να μπορέσουμε ε, να αξιολογήσουμε την πρόοδο προ συστήματα βιώσιμα, συνταξιοδοτικά συστήματα βιώσιμα, η Επιτροπή έχει ε, θέσει στην Επιτροπή ε, Κοινωνικής Προστασίας κάποιους δείκτε και αυτά θα χρησιμοποιηθούν και στο πλαίσιο τη Στρατηγική για την Ευρώπη 2020 για να και της κοινωνικής προστασίας και των συνταξιοδοτικών συστημάτων στα κράτη-μέλη. Η συνταξιδοτική μεταρρύθμιση πρέπει να βασίζεται σε λύσεις που θα διατηρούν την επάρκεια και την βιωσιμότητα των συντάξεων και όχι εις βάρος των ηλικιωμένων και των περισσότερο ευάλωτων από κοινωνική πλευρά. Στις πολιτικές κατηστήρες γραμμές το Σεπτέμβριο ο πρόεδρος Μπαρόζο είπε ότι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι συντάξεις ε, θα πληρούν το ρόλο που έχουν, δηλαδή το να δώσουν την μέγιστη υποστηρίξη στους ε, συνταξιούχους και τώρα και στο μέλλον και ιδίω στι ευάλωτε ομάδε. Επαρκή συντάξη επομένω, σημαίνει ότι δεν θα, δεν θα διατρέχουν τον κίνδυνο τη φτώχεια οι πολίτε και θα μπορούν να διατηρήσουν ένα επίπεδο διαβίωση ε, σε ένα λογικό βαθμό μετά τη συνταξιοδότησή του. Δεδομένη τη τωρινή πίεση στα συστήματα συνταξιοδότηση και δεδομένων των προβλημάτων για τι εναλλακτικέ λύσει, όπω είναι οι υψηλότεροι φόροι ή οι συμπληρωματικέ εισφορέ για του πιο φτωχού συνταξιούχου, καταλαβαίνουμε όλοι ότι ε, για τη διασφάλιση των συντάξεων ε, ώστε να είναι βιώσιμες ε, και επαρκείς θα χρειαστεί μεγαλύτερος χρόνος εργασίας. Η Επιτροπή δεν μπορεί από μόνη της να τα επιτύχει όλα θα πρέπει και οι εργαζόμενοι να καταλάβουν ότι θα πρέπει να εργάζονται περισσότερο για να μπορούν να έχουν αυτά τα δικαιώματα συνταξιοδότηση. Αυτό σημαίνει ε, ανοιχτή αγορά εργασίας, παροχή κατάρτισης ε, και ενημέρωσης των δεξιοτήτων τους καθ' όλη τη ε, διάρκεια της των χρόνων εργασίας τους και διασφάλιση της βελτίωσης των συνθήκων υγείας και υγιεινής. Η Στρατηγική Ευρώπη 2020 αποτελεί το γενικότερο πλαίσιο για τις προσπάθειες αυτές που πρέπει να καταβληθούν. Τα κράτη-μέλη έχουν θέσει ψηλά τον πύχη στα πρώτα προγράμματα ε, της μεταρρύθμισης και το τωρινό ευρωπαϊκό πλαίσιο για της συντάξεις θα πρέπει να ενημερωθεί στο πλαίσιο των δημογραφικών αλλαγών και των διδαγμάτων βάσει της περίοδου κρίσης που διανύουμε και αλλαγών στα συνταξιοδοτικά προγράμματα. Η πράσινη βίβλος για το συνταξιοδοτικό ανοίγει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη μελλοντική συζήτηση μετά την υιοθέτησή του τον Ιούλιο, ούτως ώστε να διαμορφωθεί ένα σύστημα συντάξεων με ασφάλεια και αξιοπιστία. Η πράσινη βίβλος καταγράφει ότι είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών το συνταξιδοτικό σύστημα, αλλά παράλληλα προσπαθεί να συνεισφέρει στην προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωση για τα συνταξιδοτικά συστήματα. Προσπαθεί να εξετάσει πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει τα κράτη-μέλη, ώστε να διαμορφώσουν ε, συνταξιδοτικά συστήματα επαρκή και βιώσιμα στο μέλλον, ώστε να είναι αυτά τα συστήματα ισχυρά. Η Πράσινη Βίβλος ε, ενδιαφέρει ε, και τα κράτη-μέλη και τους εργοδότες ε, και τα συνδικάτα που παίζουν ρόλο κλειδί σε ορισμένα συνταξιοδοτικά συστήματα και βέβαια ενδιαφέρει και άμεσα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όλα μας τα μέτρα θα πρέπει να βασιστούν σε τεκμήρια τα οποία θα έχουμε διαπιστώσει και θα τηρούν πλήρως τις αρχές της επικουρικότητας. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Μπλίνκεβιτσιούτε, αλλά όχι σε συμπληρωματικέ ερωτήσει, ε, γιατί ήταν αρκετά μακροσκελή η απάντηση του Επιτρόπου. Κυρία Μπλίνκεβιτσιούτε. Σα ευχαριστώ για την απάντηση, κύριε Επίτροπε. Αυτό που θα ήθελα να ακούσω από εσά όμω είναι ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την απασχόληση των ηλικιωμένων, διότι η πράσινη βίβλος στην οποία αναφέρατε δηλώνει ότι θα πρέπει η ηλικία συνταξιοδότησης ε, να μεταφερθεί ε, βάσει των δημογραφικών αλλαγών και της γύρωσης του πληθυσμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να δούμε όμως πώς φύγονται οι πολίτες από αυτή την ε, επιμήκυνση του χρόνου εργασίας. Κύριε Επιτροπέ, έχετε το λόγο και παρακαλώ να είστε σύντομος. Ένα από τα βασικά μέτρα που ακολουθούν την εργασία μας για τις συντάξεις είναι η Ευρωπαϊκή Χρονιά του 2012 η οποία βρίσκεται σε στάδιο προετοιμασίας. Θα υπάρξουν προπαρασκευαστικές δημογραφικές εργασίες έτσι ώστε να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξει και τις δυνατότητες απασχόλησης των ηλικιωμένων, των μεγαλύτερων σε ηλικία, ιδιαίτερα μέσω του προγράμματος διαβίου κατάρτισης και μέσω της διατήρησης φυσικά της υγείας των εργαζομένων. Το επόμενο θέμα είναι το θέμα του κυρίου Παπανικολάου. Είναι η ερώτηση υπαριθμή Ε, για τον κύριο Κρόουλη μπορεί να προετοιμάσει μια συμπληρωματική για την οίκοση του κύριου Παπα-Νικολάου. Λοιπόν, Επίτροπε, ε, απάντηση στο θέμα των επιπτώσεων των νέων εργασιακών σχέσεων ε, για την νεολαία και συμπληρωματική ερώτηση του κυρίου Κράουλη για την ανική ανεργία γενικότερα. Το μνημόνιο το οποίο υπέγραψαν ε, οι αρχές οι ελληνικές με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λέγει ότι η Ευρωπαϊκή ε, κυβέρνηση θα πρέπει να νομοθετήσει για συγκεκριμένες ομάδες και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας όπως οι νέοι. Υπάρχουν ομάδες λοιπόν οι οποίες αντιμετωπίζουν υψηλά, ε, υψηλούς κινδύνους ανεργίας και κινδύνους αποκλεισμού. Πολύ συχνά πληρώνονται και σε άλλα κράτη-μέλη όπως το Βέλγιο, την Τσεχία, τη Γαλλία, τη Μάλτα, την Ολλανδία, τη Σλοβακία και την Πορτογαλία λιγότερα οι νέοι. Το βασικό επιχείρημα για τον ελάχιστο μεστό είναι να καταπολεμηθεί φυσικά η φτώχεια αλλά παρόλα αυτά οι μισθοί μερικές φορές αυξάνουν το κόστος εργασίας και μπορούν να παρεμποδίζουν την είσοδο των νέων στην αγορά εργασίας. Το υψηλό ποσοστό ανεργίας ανάμεσα στους νέους στην Ελλάδα αποδεικνύει την δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι νέοι για να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Από τους 15 μέχρι τα 29 φτάνουμε σε ένα ποσοστό ανεργίας σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία γύρω στο 30,8%. Και φαίνεται ότι η κατάσταση δεν θα βελτιωθεί άμεσα. Γενικότερα η ανεργία είναι υψηλή στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στον τομέα της μακροπρόθεσμης ανεργίας. Κάποια μέτρα στο Μνημόνιο Συνεργασίας και Κατανόησης προβλέπουν τον καθορισμό ονομαστικών επιπέδων αμοιβών για μία περίοδο τριών ετών για αυτούς οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα εισόδου στην αγορά εργασίας όπως οι νέοι και οι μακροπρόθεσμα άνεργοι. Φυσικά η ποιότητα των θέσεων αυτών απασχόλησης είναι βασικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ακριβώς προβλέπεται και φάνηκε και από την προηγούμενη συζήτηση. Συστηματικά προσπαθούμε να προτείνουμε μέτρα για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και να προωθήσουμε την κοινωνική συνοχή. Τα μέτρα αυτά υποστηρίζονται από το Κοινωνικό Ταμείο κυρίως και από άλλα ταμεία το Κοινωνικό Ταμείο στην Ελλάδα χρηματοδοτεί πολλά μέτρα για να βοηθήσει την ένταξη στην αγορά εργασίας νέους, γυναίκες και μακροπρόθεσμα ανέργους. Πάρα πολλά μέτρα όπως είπα, όπως ε, προσωπικές υπηρεσίες προς τους ανέργους, κάλυψη των αναγκών των ανέργων, προώθηση της απασχολησιμότητά τους, βελτίωση των ικανοτήτων τους, βελτίωση της κοινοτικότητάς τους κτλ. Το Μνημόνιο Συνεργασίας θέτει στόχους για την Ελλάδα λοιπόν για να βελτιώσει την χρήση των διαφθορτικών ταμείων και να οδηγηθεί σε υψηλότερη απασχόληση και οικονομική ανάπτυξη. Μισό λεπτό ο κύριος Παπα-Νικολάου και μισό λεπτό μετά ο κύριος Κράουλη. Συγγνώμη αλλά δεν θα δώσω το λόγο σε άλλον. Κύριος Παπα-Νικολάου έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε για την απάντησή σας. Δεν κατάλαβα βεβαίως αν όσα προβλέπονται στο μνημόνιο είναι τελικά προτάσεις της Επιτροπής ή και σκέψεις ελληνικής κυβέρνησης που κατέληξαν τελικά σε αυτά τα συμπεράσματα σε σχέση με, το μειωμένο, ε, με τις μειωμένες απολαβές που πρέπει να έχουν οι νέοι εργαζόμενοι. Στο μνημόνιο προβλέπετε επίσης, και αναφέρατε κι εσείς κάποια νούμερα, ότι μέχρι το 2012 η ανεργία θα βαίνει αυξανόμενα σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, με πιο ευάλωτη αυτή των ηλικιών 20 με 25 ετών. Και ρωτώ, πώς θα φτάσουμε στο 2020 και θα προσεγγίσουμε τους στόχους των στρατηγικών μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έστω και σε κάποιο

προς την Επιτροπή, συγκεκριμένα προς τον Επίτροπο, θα ήθελα να πω ότι λόγω των προκλήσεων που ε, αντιμετωπίζουν οι νέοι στην κατάρτιση και την απασχόληση, απαιτούνται νέες πρωτοβουλίες, ακριβώς στοχευμένες προς αυτή την ομάδα για να βρεθούν οι κατάλληλοι τρόποι. Και ένα από τα σημεία που δεν βλέπω στις προτάσεις της Επιτροπής είναι η χρήση του διαδικτύου και των κοινωνικών δικτύων ε, για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε τους νέους ε, ώστε να κάνουν αίτηση για κατάρτιση ή να προβάλλουν τις απόψεις τους. Έχουν, έχει κάποιες ιδέες η Επιτροπή από αυτού. Κύριε Επίτροπε, όχι πάνω από δύο λεπτά παρακαλώ. Χωρί μικρόφωνο. Χωρίς μικρόφωνο, Επίτροπο. Oh, sorry. So, uh, I would like to just refer to the θα αναφερθώ στην πρωινή ομιλία του Προέδρου της Επιτροπής όπου παρέθεσε ορισμένες ιδέες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και για την κινητικότητα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς αυτά μπορούν να ενισχυθούν, ιδίως προς όφελος των νέων. Υπάρχουν αρκετά προγράμματα επ' αυτού και θα ήθελα ε, να μιλήσω για την ε, πρόταση της επόμενης εβδομάδας για την κινητικότητα των νέων που συνδυάζει πρωτοβουλίες ε, για ευκαιρίες απασχόλησης για τους νέους, όχι συγκεκριμένα στην Ελλάδα, αλλά είμαι βέβαιος ότι και η Ελλάδα θα υποφεληθεί από την ε, προσπάθεια αυτή. Ευχαριστώ. Thank you. Uh, Mr. Crowley, of course, your question. Ευχαριστούμε. Θα απαντηθεί εγγράφως η ερώτησή σας, ε, κύριε Κράουλη. Θα λάβετε πλήρη απάντηση. Ο κύριος ε, Πατεκόπ Γκάλεχερ δεν είναι εδώ. Επομένως, περνάμε στην ερώτηση 23, Μίτσελ, για τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας και τη διάσκεψη κορυφής ερώτηση η οποία απευθύνεται στον Επίτροπο Πίμπαλξ. Θα περιμένουμε να εγκατασταθεί για να ακούσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον την σύντομη απάντησή του. Ευχαριστώ πολύ Πέντε χρόνια μένουν μόνο για να επιτευχθούν οι αναπτυξιακοί στόχοι τη ε, χιλιετίας. Ε, ο στόχος ήταν το 2015 και η Επιτροπή εξακολουθεί να πιστεύει ότι είναι εφικτό ο στόχος αυτό όπως και οι άλλοι εταίροι, δείχνουμε ισχυρή ε, πολιτική δέσμευση για την εφαρμογή των απαραίτητων πολιτικών και θα πρέπει να λάβουμε συγκεκριμένη δράση με βάση τα διδάγματα που έχουμε αντιλήσει. Πολλές ε, χώρες έχουν ε, σημειώσει σημαντική πρόοδο για την επίτευξη των στόχων και φαίνεται ότι θα τους επιτύχουν. Κάποιε άλλε χώρε όμω ενδέχεται να αντιμετωπίσουν δυσκολίε. Η συνεδρία της Ολομέλη του του 2010 πράγματι αντιπροσωπεύει μια πρόκληση. Ωστόσο, ο στόχος της Κομισιόν δεν είναι μόνο να επιβεβαιωθούν οι δεσμεύσει που αναλήφθηκαν το 2000. Στόχος τη επιτροπή είναι να έχουμε ένα απτό αποτέλεσμα που θα ε, οδηγήσει στην εκπλήρωση των στόχων του 2015 για το μέλλον. Η επίτευξη των στόχων της χιλιετίας αποτελούν πρώτα απ' όλα υποχρέωση της κάθε μεμονωμένης χώρας. Ό,τι αφορά τη διεθνή υποστήριξη, την ε, διεθνή χορήγηση βοήθειας, η ευρωπαϊκή κοινότητα είναι ένας από τους σημαντικότερους χρηματοδότες ε, και αποτελεί ένα καλό παράδειγμα για τους εταίρους. Της βάση προτάσεων της Κομισιόν, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν μία δέσμη φιλόδοξων και συγκεκριμένων δράσεων και πολιτικών μέχρι το 2015. Και αυτή η δέσμη είναι μια κοινή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν ναι, και της διάσκεψης κορυφής και επέκεινα των, ε, της διάσκεψης κορυφής των Ηνωμένων ε, Εθνών. Το συμπέρασμα του Ιουνίου νομίζω ότι εκφράζει τη δέσμευσή μας για την επίτευξη των στόχων και τα κράτη-μέλη συμφώνησαν ε, σε αιτήσια αξιολόγηση της προόδου με βάση τη σχετικής, ε, βάση της σχετικής έκθεσης του Συμβουλίου. Ελπίζουμε να γίνει κάτι αντίστοιχο σε τέτοια βάση και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στη διάσκεψη κορυφής του Σεπτεμβρίου επαναλαμβάνουμε τη δέσμευσή μας. Στόχος είναι όχι το 0,7 του ΑΕΠ για την Απτυξιακή βοήθεια μέχρι το 2015. Ευχαριστώ κύριο Μίτσελ. Θέλω να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για την απάντησή του σε αυτού του δύσκολου καιρούς. Συμφωνεί η Κομισιόν μαζί μου ότι είναι απαραίτητο να ενημερώνουμε την κοινή γνώμη για τις επιτυχίε που έχουμε σε ό,τι αφορά τον αναπτυξιακό προπολογισμό που δαπανούμε. Και δεύτερον, συμφωνείτε με την μείωση αυτή του ΑΕ. Ίσως ε, δεν θα έπρεπε να μειωθεί το ποσοστό του μειωμένου ακαθάριστου εθνικού εισοδήματο. Η δημόσια υποστήριξη σίγουρα είναι πολύ σημαντική, λέει ο επίτροπο, επομένω εξίσου σημαντική είναι η πληροφόρηση προβολή και επομένως έχουμε αναλάβει ω Επιτροπή διάφορα προγράμματα τις ε, μέρε αυτής για την ανάπτυξη και θα αναφέρουμε ό,τι έχουμε επιτύχει και θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια. Ό,τι αφορά ε, τη μείωση του εισοδήματος πράγματι με τη μείωση ε, θα έχουμε μείωση σε κάποιες χώρες αλλά και πάλι είμαστε γύρω στο 0,4%. 100. Πρέπει λοιπόν να δουλέψουμε σκληρά για να φτάσουμε στο 0,7% και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζω ότι δεν θα πρέπει να αυξηθούν τα ποσά ούτε σε σχετικές τιμέ ούτε σε απόλυτε τιμέ, γιατί είμαστε χαμηλότερα από τις δεσμεύσεις που αναλάβαμε και η αξιοπιστία μας εξαρτάται ακριβώς από το επίπεδο και των δεσμεύσεων που αναλαμβάνουμε και των αποτελεσμάτων που φέρνουμε σε ό,τι αφορά την ε, επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας. Ήρθε ο κύριος Γκάλαχερ τώρα. Θα μπορούσατε να απαντήσετε λοιπόν την ερώτηση 22 για την επικείμενη διάσκεψη Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής. number 22, yeah. Just a second. <laughs> Uh, well, uh, the political issues to... forthcoming uh, EU-Africa summit. Τα πολιτικά ζητήματα που θα αντιμετωπιστούν στην επικείμενη διάσκεψη Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής συζητώνται μαζί με άλλα θέματα που συζητούμε παρόμοιους φορείς σύμφωνα και με τα συμπέρασματα που εξάγονται από τη συνθήκη της Λισαβόνας και η Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα η Επιτροπή ε, θα παίξει ρόλο κλειδί μέσα σε αυτή την επικείμενη διάσκεψη η διάσκεψη η οποία θα γίνει το, στη Λιβύη στο τέλος Νοεμβρίου 2010 θα ορίσει με πιο συγκεκριμένο ε, τρόπο το πεδίο συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικής κατά τα προσεχή έτη. Ιδίω η διάσκεψη κορυφή θα πρέπει να συμφωνήσει για τις νέες μεθόδους εργασίας τις του νέου κοινού προγράμματος δράσης για τη Στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση Αφρικής για τα έτη 2011-2013. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η στρατηγική της Λισαβόνας το 2007 και η διάσκεψη κορυφή τη Λισαβόνα ε, ασχολήθηκε με την αναβάθμιση ε, του ρόλου αυτής της διάσκεψης Και το 2010 η διάσκεψη θα πρέπει ε, να ασχοληθεί με την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων. Η Επιτροπή θέλει στη διάσκεψη κορυφής ε, να ασχοληθούν ε, τα εξή θέματα. Δημιουργία θέσεις απασχόληση, θέσεων απασχόλησης ε, και επενδύσεων. που θα μας δώσει τη δυνατότητα να έχουμε οικονομική ανάπτυξη και βελτίωση των τομέων όπως η ενέργεια, η ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, το εμπόριο, αλλά και η γεωργία και η ασφάλεια των τροφίμων. Η περιβαλλοντική προστασία και ιδίως εστιάζοντας στην βιοπικιλότητα και στην κλιματική αλλαγή θα είναι ένα από τα σημαντικά θέματα. Ακόμη η ειρήνη και η ασφάλεια, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της πειρατείας και η καταπολέμηση ε, της ε, διαμεθοριακής εγκληματικότητας. Αυτά συνδέονται και με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Επιτροπή ε, προσδοκά ότι πολλοί ηγέτε από τις γειτονικέ χώρες ε, θα παρευρεθούν σε αυτή τη διάσκεψη κορυφή. και περιμένουμε ότι τα αποτελέσματα θα φτάσουν ε, σε ευρία κλίμακα σε πολλούς ενδιαφερομένους από ολόκληρο τον κόσμο και θα ευλακούν επίσης και τα κοινοβούλια και η κοινωνία των πολιτών. Ακόμη η Επιτροπή θέλει να συμμετέχουν και άλλοι εκπρόσωποι από διάφορους φορείς στην Αφρική, από πανεπιστήμια, από ερευνητικούς φορείς, από οργανώσεις νέων και από τοπικές αρχές. Όπως και στην προηγούμενη διάσκεψη κορυφής, και αυτή η διάσκεψη κορυφή ε, θα καταλήξει τελικά σε πολιτικέ δηλώσει υψηλού επίπεδου ή και σε κοινέ δηλώσει αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Γκάλεγερ. Μισό λεπτό. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και τον Επίτροπο που απάντησε στην ερώτησή μου. Είναι πολύ σημαντική αυτή η διάσκεψη κορυφής και χαίρομαι που πληροφορούμε από τον Επίτροπο σχετικά με τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν, όπου θα συμπεριλαμβάνουν την ανάπτυξη, τις θέσεις απασχόλησης, το περιβάλλον, την ειρήνη και την ασφάλεια. Είναι επίσης σημαντικό ότι μας είπε ότι θα υπάρχουν και συγκεκριμένα παραδοτέα, συγκεκριμένα αποτελέσματα τα οποία αναμένουμε. Και είναι σημαντικό να σας ζητήσω κύριε Επίτροπε να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες που έχετε ούτως ώστε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κατανοήσουν τη σημασία της αναπτυξιακής βοήθειας και να κατανοήσουν τα κράτη-μέλη ότι τώρα σε μια εποχή ύφεσης θα πρέπει να μην μειώσουμε την αναπτυξιακή βοήθεια. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, αν μπορείτε σύντομα. Πραγματικά η δική μου δουλειά είναι να ενθαρρύνω τα κράτη-μέλη να ε, ε, ενισχύσουν την αναπτυξιακή τους βοήθεια και είμαστε υπερήφανοι γιατί είμαστε οι μεγαλύτεροι δωρητές. Διαφορετικά θα, θα υπήρχε μεγαλύτερη αστάθεια στον κόσμο και μεγαλύτερη φτώχεια. Χάρη στη δική μας βοήθεια υπάρχουν τα καλά αποτελέσματα όπως ανέφερε και ο πρόεδρος ε, του Μάλι σήμερα το πρωί, το μεσημέρι κατά τη δήλωσή του ενώπιον της Ολομέλειας. Ευχαριστώ πολύ. Μόνο ε, Δύο ερωτήσεις θα απαντηθούν όπω είπα στην αρχή και γι' αυτό στον κύριο Πόσελ και στην Βαρόνη θα δοθούν γραπτό οι ερωτήσει. Και περνώ ε, στις ερωτήσεις προς την κυρία Χέντεγκαρντ. Πρώτη ερώτηση από την κυρία Τικάου, η ερώτηση υπαριθμών 26. Σας παρακαλώ όμως να είστε πολύ σύντομοι προς όλους τους συναδέλφους. Κύριε Χέντεγκαρντ, έχετε το λόγο. Thank you very much. Το 2007 και στις αρχές του... 2006 και αρχές 2007 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει μια μελέτη για τα φαινόμενα ξηρασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά από την αξιολόγηση αυτή παρουσίασε κάποιες πολιτικές δυνατότητες επιλογής έτσι ώστε να εξοικονομηθεί η κατανάλωση υδάτων Αυτό δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2007. Επτά ε, επιλογές πολιτικής ε, εντοπίστηκαν και σχεδιάστηκαν για την καταπολέμηση του προβλήματος της ξηρασίας. Πρώτον, σωστή τιμολόγηση των υδάτινων πόρων, καλύτερη χρηματοδότηση των υποδομών, διαχείριση κινδύνου, βελτιωμένη διαχείριση κινδύνου, βελτίωση των πρακτικών, ενίσχυση της ε, κουλτούρας και της νοοτροπίας εξοικονόμησης ύδατος και επίσης επεξεργασία των λιμάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν προετοιμάζει ετήσιες εκθέσεις που αξιολογούν την εφαρμογή αυτών των πολιτικών επιλογών στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφαρμόζει το Λευκό Βιβλίο για την καταπολέμηση των κλιματολογικών αλλαγών, των συνεπειών των κλιματολογικών αλλαγών και η ένταξη αυτών των στοιχείων στις μείζονες κοινοτικές πολιτικές θα γίνει ήδη από τον επόμενο χρόνο. Το 2012 θα υπάρξει μια ανακοίνωση επίσημη για την κατάσταση των υδάτινων πόρων όπως επίσης και ε, το κατά πόσον επηρεάζονται από τις κλιματολογικές αλλαγές η κατάσταση των υδάτινων πόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προωθούμε πιλωτικά προγράμματα για να αντιμετωπίσουμε την απερίμωση ή ερημοποίηση στην Ευρώπη και να ενισχύσουμε τους υδάτινους πόρους απέναντι στις κλιματολογικές αλλαγές. Η ξηρασία και η απερίμωση αντιμετωπίζονται επίσης και από τομεακές πολιτικές όπως ε, ανάπτυξη της υπαίθρου στα πλαίσια της ΚΑΠ και πολιτικές συνοχής φυσικά. Ευχαριστώ η κυρία Τικάου μισό λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Επίτροπε, η καταπολέμηση των κλιματολογικών αλλαγών, των συνεπειών των κλιματολογικών αλλαγών είναι μια προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι επιπτώσεις των κλιματολογικών αλλαγών είναι ορατές όλο και περισσότερο. Γι' αυτό λοιπόν τι θα κάνει έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντικατοπτρίζει το πρόβλημα αυτό και πώς θα χρησιμοποιήσετε τα πολιετή χρηματοδοτικά προγράμματα για να καλύψετε τις ανάγκες στο συγκεκριμένο τομέα. Ευχαριστώ λέει η Επίτροπος Χέντεγκαρντ. Ήδη από τον Ιανουάριο είχαμε πει ότι θα προσπαθήσουμε στα πλαίσια των νέων δημοσιονομικών προοπτικών να ελέγχουμε κλιματολογικά τις πολιτικές μας και τα προγράμματα. Εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση, σαν παράδειγμα, χρηματοδοτεί μια μεγάλη υποδομή, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να βλέπουμε ήδη στην φάση της κατασκευής να λάβουμε υπόψη μας την γνώση την οποία έχουμε για τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιστεί το θέμα των υδάτων και το γενικότερο πρόβλημα του κλίματος. Προσπαθούμε λοιπόν εμείς να ελέγξουμε κλιματολογικά τον τρόπο με τον οποίο θα πανούμε γενικότερα χρήματα και επενδύουμε και να υποστηρίξουμε οικονομικά προγράμματα μόνο τα οποία σίγουρα αποδεικνύεται ότι μπορούν να επωφεληθούν από τις γνώσεις που έχουμε για τους συγκεκριμένους τομείς. Είναι ένα συγκεκριμένο, αν θέλετε, παράδειγμα. Right. Καλώς. Περνάμε τώρα στην 27 και 28. Φλόρεντς και Ροντρίγες. Έχετε το λόγο, Επίτροπε. Σας ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω, ναι, όπως είπατε, να απαντήσω από κοινού και τις δύο ερωτήσεις αφορούν και οι δύο ότι η στρατηγική μέχρι το Κανκούν και νομίζω ότι στους ε, εδώ παρόντες είναι γνωστό ότι ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αλλαγή του κλίματος είναι ένας ε, συνολικός ε, στόχος για μια συνολική νομικά δεσμευτική ε, συμφωνία ώστε να μην αυξηθεί η θερμοκρασία του πλανήτη πάνω από δύο βαθμούς. Βέβαια θα πρέπει αυτή η συμφωνία να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατόν. Αυτό υποστηρίζαμε στην Κοπενχάγη, αυτό εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε. Είμαστε έτοιμοι να ε, υποστηρίξουμε την ε, σχετική αυτή πρόταση και στο Κανκούν τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο. Θα πρέπει πάντως να αναγνωρίσουμε ότι για μια ακόμη φορά υπάρχουν άλλοι οι οποίοι μάλλον δεν θα είναι έτοιμοι την προηγούμενη εβδομάδα σε μια υπουργική διάσκεψη αυτό συζητήθηκε. Μάλλον έτσι θα έχουν τα πράγματα. Πρέπει λοιπόν να είμαστε ρεαλιστές. Και νομίζω ότι βήμα-βήμα η σταδιακή αυτή προσέγγιση που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Μάρτιο ε, και υποστηρίζεται αυτή η πολιτική. Αυτό λοιπόν επιδιώκουμε αυτή τη στιγμή, να πάμε βήμα-βήμα. Ποιο είναι το μείζον ζήτημα τι μπορούμε να επιτύχουμε, τι είδου δέσμη μπορεί να εγκριθεί στον Κανκούν. Κατά την άποψή μας θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε βασικά ζητήματα αρχιτεκτονικής και να δρομολογήσουμε μείζονε δράσεις ε, με βάση μια δέσμη αποφάσεων. Και θα μπορούσε αυτή η δέσμη αποφάσεων στο Κανκούν να περιλαμβάνει τα εξή στοιχεία. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να βασιστούμε και να εκμεταλλευτούμε τα ε, ζητήματα που έχουμε ήδη αποφασίσει και αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίσουμε στο Κανκούν με την υιοθέτηση συγκεκριμένων αποφάσεων. Θα πρέπει επίσης και είναι πολύ σημαντικό να γίνει σημαντική πρόοδο σε ό,τι αφορά τη μέτρηση, την αναφορά και την επαλήθευση της μείωσης των εκπομπών και την οικονομική στήριξη. Αυτό είναι επίσης σημαντικό στοιχείο η απερίμωση, η αποψήλωση των δασών μάλλον, μείωση των εκπομπών, μηχανισμοί αποψήλωση των δασών, υποβάθμιση των δασών, αυτό ε, το συστήσαμε στην Κοπενχάγη και θα πρέπει να είναι και ένα από τα παραδοτέα αποτελέσματα μια δέσμη ε, που θα εγκριθεί στο Κανκούν. Είμαστε πολύ κοντά να το συμφωνήσουμε στην Κοπενχάγη. Νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε μια φιλόδεξη απόφαση για την ε, δασοκομεία. Το ίδιο θα πρέπει να γίνει σε ό,τι αφορά το πλαίσιο για δράση και προσαρμογή και για την τεχνολογία και την τεχνολογία τεχνολογική συνεργασία θα δούμε κατά πόσο θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν κάποια μέτρα στις αποφάσεις του Κανκούν. Επίσης θέλουμε να έχουμε σημαντική πρόοδο στην οικονομική αρχιτεκτονική. Δεν χρειάζεται καν να πω ότι σε ό,τι αφορά την ταχεία χρηματοδότηση Υπάρχουν σημαντικά ζητήματα και ένα από αυτά στο Κανκούν θα είναι κατά πόσον ο υπόλοιπο κόσμο ε, θα θέλει να τηρήσουν τι δεσμεύσει του ε, και ανεψόμενε χώρε. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να συζητήσουμε και την αρχιτεκτονική ε, για τη μακροπρόθεσμη στρατηγική και για ένα ταμείο για την κλιματική αλλαγή. Θα θέλαμε να υπάρχουν αλλαγές για τη νέα αγορά άνθρακα, να δούμε αν θα μπορούσαμε να προωθήσουμε τα συστήματα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών και βέβαια και έχουμε και εμείς ένα ευχολόγιο που αφορά τις εκπομπές ε, από τις αεροπορικές και τις θαλάσσιες μεταφορές. Σε ό,τι αφορά τις, ε, το μετριασμό και τις ασμές που έχουν αναλυφθεί, πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνουν και εκεί κάποια πράγματα αν καταφέρουμε στο Κανκούν θα έχουμε ένα διεθνές πλαίσιο και αν έχουμε συμφωνήσει επί της ουσίας ίσως ε, την επόμενη φορά θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε και με μια πιο σαφή νομική μορφή κάποια πράγματα. Η έκβαση στο Κανκούν πάντως πρέπει να είναι ισορροπημένη και τι εννοώ με τη λέξη ισορροπημένη. Το πρωτόκολλο του Κιώτο υπό την τρέχουσα μορφή του δεν μπορεί από μόνο του να επιτύχει το στόχο του να μείνουμε κάτω από την αύξηση θερμοκρασία κάτω των δύο βαθμών. Ναι, λοιπόν, είμαστε ανοιχτοί σε μια δεύτερη περίοδο δέσμευση. Αλλά θα πρέπει να είναι σαφές προς όλους ότι αυτό από μόνο του δεν αλλάζει και πολλά πράγματα. Πρέπει να υπάρξουν και κάποιε προποθέσει. Αλλιώ εμεί θα είναι δύσκολο να πιέσουμε άλλου ε, να, κάνουν, να αναλάβουν δεσμεύσεις στο μέλλον. Θα πρέπει να επιδιώξουμε συγκρίσιμε δεσμεύσει ε, με άλλε χώρε ε, που δεν είναι συμβαλόμενα μέρη στο πρωτόκολλο του Κιώτο, όπω είπα φυσικά. Και θα πρέπει να έχουμε κάποιε δράσει και με μείζονε αναδυόμενες οικονομίε, όπω στην Κίνα για παράδειγμα. Υπάρχουν όμω και άλλοι όροι και προϋποθέσεις που θα πρέπει να έχουμε εκπληρώσει κατά κάποιο τρόπο ώστε να έχουμε αυτή τη δεύτερη περίοδο. Μιλώ για την περιβαλλοντική ακαιρεότητα. Σήμερα υπάρχουν κάποιες αδυναμίες στο πρωτόκολλο του Κιώτο και αυτές ε, υπονομεύουν την περιβαλλοντική ακαιρεότητα. Θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε αυτά τα αδυνατά σημεία. Ειδικότερα σε σχέση την δασοπονία, τη δασοκομεία και το AAUs για τις εκπομπές. Αν δεν καταφέρουμε πρόοδο σε αυτού του τομεί, δεν θα καταφέρουμε να μειώσουμε την αύξηση τη θερμοκρασία κάτω των δύο βαθμών. Σήμερα απαγορεύουν οι κανόνες του Κιώτο η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να καλύπτει κάτι εκπομπές από την αεροπορία και έχουμε και το σύστημα CDM Όλα αυτά θα πρέπει να αλλάξουν στη μελλοντική διάταξη και έτσι μόνο θα μπορέσουμε να έχουμε αυτή τη δεύτερη περίοδο δέσμευση. Αλλιώ δεν θα την καταφέρουμε. Θα πρέπει να πω επίση ότι υπάρχει έλλειψη ισορροπία στι διαπραγματεύσει. Η διαπραγματεύσει για τη συνέχιση του Κιώτο είναι πολύ πιο προηγμένες και προχωρημένες σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις για τις νέες δράσεις με τις ΗΠΑ και τις αναπτυσσόμενες χώρες. Και θα πρέπει να έχουμε στη δεύτερη περίπτωση σημαντική πρόοδο αν θέλουμε να επιτύχει το Κανκούν. Και αν δεν θέλουμε να πάμε εκεί απλά για να είμαστε εκεί και όχι για να σημειώσουμε σημαντική πρόοδο. Για να υπάρξει επιτυχία λοιπόν στο Κανκούν θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να ηγείται δίνοντα το καλό παράδειγμα. Είμαστε ηγέτε ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή, είμαστε στη σωστή πορεία, θέλουμε τη μείωση του 20%, την έχουμε κάνει νόμο και θα αυξήσουμε το στόχους μας στο 30% εάν υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Επίσης, ό,τι αφορά την ε, ταχεία χρηματοδότηση, το fast track financing, επίσης τα πάμε καλά, αλλά δεν είμαστε εμεί το πρόβλημα. Και το τελευταίο, διεξάγουμε, μάλλον προσπαθούμε να προσεγγίσουμε πολλές άλλες χώρες και μαζί με τις διπλωματικές υπηρεσίες του Συμβουλίου προσπαθούμε να δρομολογήσουμε ένα δίκτυο πράσινης διπλωματίας μέχρι το Κανκούν. Στόχος μας είναι να ευαισθητοποιήσουμε τους χαράκτε πολιτικών αποφάσεων, να τους ε, προσετεριστούμε και σίγουρα θα πρέπει αυτή η καθημερινή επαφή να ενταθεί ακόμη περισσότερο μέσω του δικτύου των αντιπροσωπιών. Και φυσικά θα θέλαμε και με το Κοινοβούλιο σε αυτές τις ε, δράσεις μας να συνεργαστούμε. Είχα σε μια συνάντηση με τους επικεφαλής αντιπροσωπιών ε, την δυνατότητα να το πω στους, ε, στις διάφορες αντιπροσωπείες. Ελπίζω να έχουμε μια καλή συνεργασία και καλή ανταλλαγή απόψεων για να το επιτύχουμε και να έχουμε και μια θετική, μια ισχυρότερη θέση συνολικά. Ευχαριστώ. Πολύ πλήρη και μακροσκέλη ήταν η απάντησή σα. Έχουμε δύο συμπληρωματικέ ερωτήσει και μετά σύντομη απάντηση από την Επίτροπο, γιατί στι 8.30 πρέπει να σταματήσουμε. Οπότε δυστυχώ ε, η τελευταία ερώτηση θα υποβληθεί, ε, η απάντηση τελευταία ερώτηση θα είναι έγγραφη. Ο κ. Φλόρεντ, ευχαριστώ πολύ, Επίτροπε, για τη διπλωματική σα απάντηση. Ετοιμάζουμε το ψήφισμά μα για το Κανκούν και θα πρέπει στο τέλος όταν ε, θα έχω, και αν θέλουμε να καταλήξουμε σε σαφή αποτελέσματα, να ξέρουμε τι θέλουμε. Λέτε ότι προσφέρετε το 20% ε, ενώ ο στόχο ήταν το 30%. Ε, τι σημαίνει αυτό σε νούμερα, θα μπορούσατε να μας το εξηγήσετε. Ποια είναι ακριβώ η επιθυμία της Επιτροπής. Ευχαριστώ κύριε Ροντρίγκε, 30 δευτερόλεπτα. Ε, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. η συγκεκριμένη απάντηση που μας δίνει η Επιτροπή είναι ότι είμαστε στην εμπροστοφυλακή και ότι θα μείνουμε στις προσπάθειες και ότι θα προσπαθούμε ε, τους άλλους να τους ε, πιέσουμε, εντάξει, συμφωνώ, αλλά αν μετά από αυτά καταφέρουμε, κύριε Επίτροπε, η ενιαία θέση να μεταφερθεί σε μία ενιαία φωνή, όχι σε 27 διαφορετικές φωνές, θα είναι και αυτό επιτυχία. Και επίση να πω ότι έχω τι ίδιε αμφιβολίε με τον κύριο Φλόρεν. Επίτροπε, δύο λεπτά παρακαλώ, όχι παραπάνω. Ε, εφόσον μου το ζητάτε, θα προσαρμοστώ, κύριε Πρόεδρε. Ε, εάν είναι όριμε οι συνθήκε, ε, είναι η απάντησή μου προ τον κύριο Φλόρεν. Και αυτό το οποίο είναι τώρα πολύ σημαντικό είναι τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση να σκεφτούν την ανακοίνωσή μας του Μαΐου και βέβαια χάρηκα που είδα ότι η Γαλλία, η Γερμανία και η Βρετανία μέσα των Υπουργών Περιβάλλοντος εκφράστηκαν ε, τον Ιούλιο σαφώς και ελπίζω ότι και τα άλλα κράτη-μέλη θα ακολουθήσουν ε, την ίδια πορεία. Δέχονται ότι δεν πρόκειται για ένα θέμα διεθνών διαπραγματεύσεων και μόνο, αλλά είναι κάτι το οποίο ε, συμφέρει και, τα, και την Ευρώπη. Και είναι κάτι το οποίο θα συνεχίσουμε να συζητάμε υπό Βελγική Προεδρία με το Βέλγιο και είναι πολύ σημαντικό το μήνυμα το οποίο θα λάβουμε και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άρα και εσείς έχετε εδώ ένα σημαντικό ρόλο να παίξετε. Και προς τον κύριο Ροντρίγκε θα ήθελα να πω ότι βεβαίως ε, συμφωνώ ότι είναι απαραίτητο να μιλάμε με μία ενιαία φωνή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μόνο μία φωνή θα ακούγεται. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ακούν ε, και όλοι οι άλλοι εταίροι σε ολόκληρο τον κόσμο αυτό το οποίο έχουν να πούν οι Ευρωπαίοι εκπρόσωποι. Το μήνυμα το οποίο θα φτάνει θα είναι το μήνυμα μιας ενιαίας γραμμής και αυτό είναι σημαντικό και θέλουμε να το διασφαλίσουμε και με την Βελγική Προεδρία και στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνουμε τη διαπραγματευτική εντολή ε, θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα προς τον έξω κόσμο γνωρίζοντας πού βρίσκονται τα όρια μας. Ε, αλλά για να το επιτύχουμε αυτό πρέπει να έχουμε και ευέλικτη διαπραγματευτική εντολή και θα πρέπει να έχουμε διαπραγματευτική ευχέρεια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και για τα αποτελέσματα που περιμένουμε από το Κανκούν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, Επίτροπε. θα στελούν απαντήσεις γραπτός για όσες ερωτήσεις δεν προλάβαμε να απαντήσουμε λόγω έλλειψης χρόνου. Τέλος της συνεδρίασης μέχρι τις 9 που θα ξαναρχίσουμε. Ευχαριστώ.